για τα οποία έχουν εγκριθεί και διανεμηθεί. Έχετε παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Εκ μέρου τη ομάδα ΕΝΕΦ θα ήθελα να ζητήσω αλλαγή τη ημερήσια διάταξη με κοινή συζήτηση για του τζιχαντιστέ. Να αντικαταστήσουμε τη συζήτηση τη Πέμπτη το πρωί. Δεν μιλάμε γι' αυτό τώρα. Δεν περάσαμε ακόμη στις αλλαγές. Τώρα όσον αφορά τα πρακτικά. Ποιο θέλει το λόγο. Για τα πρακτικά. Όχι για την ημερησία διάταξη. Τα πρακτικά τη Συνόδου τη 8η Φεβρουαρίου. Κύριε Κάρβερ, από αυτού θέλετε το λόγο ή για κάτι άλλο. Να αποφασίσουμε για τα πρακτικά. Επομένω.